Επίση, να σα ανακοινώσω ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων συνεδρίαση τη 25η Ιανουαρίου τρέχοντο έτου έλεγξε μια σειρά εντολών βάσει του κανονισμού άρθρο 3, παράγραφο 3 και 4 και προτείνει του εξή. Άντερ Κουσκέρι, Γκαρσία Στραμών, Γκαρσία Ιέρο Καραβάλο, Μακίνταερ, Μαλινόφ, Νίλσον, Βιλέλα, Σέντο Ιαλαμπάρ, Τρεματέρα, και Βάντενχολτσα. Μπρατκόφσκι, Κοσέ, Ροάτα, Στάντλερ, Κούκοβιτ, Φαντεστούκ, Μιράνο, Μάρια, Κορέα, Ζαμόρα, Ναράχο, Εσκομπάρ και Σούμπερ. Είναι κανείς κατά του ορισμού των μελών αυτών? Όχι, οπότε ε, επικυρώνεται η έγκριση. Από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.